η συνεδρίαση την Πέμπτη μετά τις ψηφοφορίες. Σε ό,τι αφορά τις πτήσεις και τα τρένα θα επηρεαστούν πιθανότατα από την απεργία όπως και οι συγκοινωνίες, οι δημόσιες. Γι' αυτό δεν είναι μπορούμε να εξασφαλίσουμε για όλους τα ίδια μεταφορικά μέσα όπως συνήθως, ωστόσο έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα ώστε να, εξασφαλιστεί, ε, να εξασφαλιστούν μεταφορικά μέσα που θα σας επιτρέψουν να φτάσετε στα σπίτια σας το ταχύτερο δυνατό. Οι αποφάσεις, οι τελικές δεν έχουν ακόμα ληφθεί, αλλά γνωρίζουμε ήδη ότι το ταλής θα λειτουργήσει κανονικά και το shuttle μεταξύ του, ανάμεσα στο Κοινοβούλιο και το σταθμό θα λειτουργήσει επίσης, αυτό είναι εξασφαλισμένο, σε ό,τι αφορά τη μεταφορά προς διάφορα αεροδρόμια στη Γαλλία, αυτό θα εξασφαλιστεί ε, από, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το Σώμα των Κοσμητόρων έχει ε, εκδώσει ένα ανακοινοθέν που αναφέρει όλα τα συμπληρωματικά μεταφορικά μέσα που θα μας επιτρέψει να παρεκκλίνουμε από τον κανόνα των 20 χιλιόμετρων. Αυτή η παρέκκληση θα επιτρέψει σε όλους να μεταβούν σε διάφορα αεροδρόμια όπως στην Ελβετία παραδείγματος χάρη. Οι υπηρεσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου δεν θα υποχρεούνται πλέον να τηρήσουν τον κανόνα των 20 χιλιόμετρων και έτσι θα μπορέσετε να διανύσετε μεγαλύτερες αποστάσεις. Η πόλη του Στρασβούργου επίσης ενημέρωσε τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για όλες τις δυνατότητες που υπάρχουν για τη μεταφορά τους. Το Προεδρείο θα συνεδριάσει 6.30 και θα δούμε για κάθε περίπτωση πώς θα εξασφαλίσουμε τη μεταφορά σας από το Στρασβούργο, από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στο Στρασβούργο, στα σπίτια σας, το ταχύτερο δυνατόν και με τον πιο αποτελεσματικό τρόπο. Αύριο θα έχετε οριστική ενημέρωση για αυτό το θέμα. Ωστόσο, εάν προκύψουν νέα στοιχεία, νέες πληροφορίες σχετικά με τις μεταφορές, την ημέρα της απεργίας, βεβαίως θα σας ενημερώσω τη Δετάρτη το πρωί. Ολοκληρώνοντας λοιπόν, Αύριο το πρωί θα έχετε μία ενημέρωση για τη μεταφορά σας και αν υπάρχουν συμπληρωματικές πληροφορίες, συμπληρωματικά στοιχεία θα σας ανακοινωθούν την Τετάρτη το πρωί. Αν η πόλη του Στρασβούργου μας ε, ενημερώσει για κάτι το καινούριο βεβαίως θα σας το γνωστοποιήσουμε αμέσως θα φροντίσουμε να ελέγχουμε την κατάσταση έτσι ώστε να μπορέσετε να γυρίσετε στα, στις πατρίδες και στα σπίτια σας το ταχύτερο δυνατό. Αυτή είναι μια πρώτη ενημέρωση. Μην ξεχνάτε ότι αύριο το πρωί και την Τετάρτη θα υπάρξουν πιθανότητα συμπληρωματικές ενημερώσεις για τις μεταφορές. Βλέπω ότι ζητήσατε το λόγο. Σας ακούω. Ευχαριστώ Πρόεδρε για αυτές τις ε, πληροφορίες. Όλοι στην Ευρώπη και ειδικότερα στο Ηνωμένο Βασίλειο Μα εκπλήσει αυτό που συμβαίνει εδώ. Ερχόμαστε εδώ στο Στρασβούργο μια φορά το μήνα. Θα μπορούσαμε απλά και μόνο να ψηφίσουμε στο... στις Εκατομμύρια ευρώ δαπανώνται κάθε χρόνο και συσσωρεύονται από χρόνο σε χρόνο. Έφτασε πλέον η στιγμή να αντιδράσουμε. Δεν πρέπει απλά και μόνο να συνεδριάζουμε εδώ. Θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας αγαπητοί συνάδελφοι στο εξής. Η παρέμβασή σας δεν εντάσσεται στην σημερινή συζήτηση. Μιλάμε για τεχνικές λεπτομέρειες, θα μας επιτρέψουν να γυρίσουμε στα σπίτια μας την Πέμπτη. Εσείς αναφερθήκατε σε ένα διαφορετικό θέμα που αφορά τη συνθήκη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν έχει καμία σχέση με τη συζήτηση που προβλέπετε να γίνει σήμερα. Ο κύριος Περόνι θέλει να πάρει το λόγο. Ένα πράγμα θα ήθελα να προσθέσω. Το Στρασβούργο έχει το πλεονέκτημα να είναι δίπλα στη Γερμανία και μπορούμε να βρούμε περισσότερες εναλλακτικές λύσεις από εδώ από ό,τι στις Βρυξέλλες. Tym kończymy dyskusję nad tym punktem. Powtarzam, będą informacje we wtorek i w środę. Dokładne informacje na ten temat. Następna sprawa